Ιανουαρίου, στον 10 Ιανουαρίου. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την κοινή συνεδρίαση που έχουμε την Επιτροπή Ανάπτυξη για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Βάσει τη διαδικασία που από κοινού επιτροπέ εκπονούν έκθεση, ε, ετοιμάζουμε από κοινού την έκθεση αυτή και θα καταλήξουμε σε κοινή συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου. Είναι μια σημαντική διαδικασία γιατί έτσι θα καθορίσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τρίτες χώρες με 90 δισεκατομμύρια περίπου από το 2021 μέχρι το 2022. που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σημερινή μας συζήτηση. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε θα δώσω το λόγο αυτής αμέσως στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την Λίντα Μακάβιν, για τα εισαγωγικά της σχόλια. Ναι, ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να πω, συνάδελφοι, είναι ότι λίγοι μήνες μας μένουν πριν από τις ευρωεκλογέ και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν λειτουργεί το μικρόφωνο, λέει η κυρία Μακάβεν. Λειτουργεί το μικρόφωνο της κυρίας Μακάβεν. Στην αίθουσα ίσως δεν ε, λειτουργεί. Εμείς ακούμε πολύ καλά την κυρία Μακάβεν στη διερμηνία. Έλεγα λοιπόν ότι θα είμαι σύντομη, ότι μας μένουν λίγοι μήνες μέχρι τις ευρωεκλογέ, ότι είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που εξετάζουμε γιατί με αυτό αποφασίζουμε το πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εξωτερική χρηματοδότηση 2021 με 2027. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε τους τέσσερις συνεισηγητές με τις πρώτες τους ιδέες. Το κύριο θέμα μας Ξέρετε ότι γίνονται συζητήσεις, αν πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό ή όχι. Το βασικό είναι η ευελιξία. Και αν υπάρχει ευελιξία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει έναν μεγάλο και σημαντικό ρόλο για την δαπάνη των κονδυλίων. Να παρακολουθούμε πού και πώς ξοδεύονται τα χρήματα. Βάσει των συνθηκών και βάσει της αναπτυξιακής ε, πολιτικής μας που θέλει να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας και προσβλέπω και εγώ στην συνεργασία με τους συναδέρφους από την ΑΦΕΤ και την Υποβιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν τέσσερις συνεισηγητές και ο πρώτος που θα πάρει το λόγο θα είναι... Ποιος? Με ποιο να ξεκινήσω? Τεπρέντα, Έγγελ, Γκέρενς. Γκέρενς. Πρώτος Σαρλ Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν βλέπω το ενδιαφέρον και την ε, συντριπτική παρουσία εδώ, ε, θα έλεγα να έχουμε καμιά εικοσαριά ε, εισηγητέ, έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα κοινό για αυτή την τόσο σοβαρή δουλειά. Τέσσερι λοιπόν συνεισηγητέ είμαστε που προσπαθήσαμε από την αρχή της προσπάθεια να συντονίσουμε την εργασία μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάτι αξιόπιστο. Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα, όμω στο τέλος διαπιστώσαμε ότι σφυριλατήσαμε μια καλή ομάδα και μπορέσαμε να δουλέψαμε καλά, προσπαθώντας να βελτιώσουμε το κείμενο το οποίο μας είχε υποβληθεί από την Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν σχετικά με το Μηχανισμό Γειτονίας Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεργασίας ε, ε, ε, είναι ένα εργαλείο το οποίο θέλει, φιλοδοξεί να ενσωματωθεί στον ε, προϋπολογισμό. Λέω φιλοδοξεί γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει ε, να γίνει μεγάλη προσπάθεια. Από πλευρά της Κομισιόν φαίνεται να είναι δεδομένο, το ίδιο και από την Κομισιόν. Στο επίπεδο του Συμβουλίου και των κρατών μελών φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε και να αγωνιστούμε για το θέμα αυτό, γιατί η παρούσα πρακτική όσον αφορά το Αναπτυξιακό ε, Ταμείο δεν δίνει την δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ασκήσει τα βασικά του δικαιώματα. Και στην ουσία η λογική είναι, για να πούμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, σε μια μεταδημοκρατική ε, λογική ε, και ε, στην ουσία δίνονται τα περισσότερα στην εταιρική σχέση με τις χώρες του Νότου. Εάν θέλουμε πραγματικά να ε, ε, ε, λειτουργήσουμε στα πλαίσια αυτού του εργαλείου και στα πλαίσια αυτής της χρηματοδότησης δημοκρατικά και αν θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικά καλό παράδειγμα και να είμαστε εντάξει με τους εταίρους μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε τα όσα προτείνονται. Όσον αφορά την ουσία, από την αρχή προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε με τρόπο ώστε το νέο αυτό εργαλείο ε, να σεβαστεί το κεκτημένο της ε, Ένωσης ε, όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και τις δράσεις της εξωτερικής πολιτικής γενικότερα. Ε, επίσης προσπαθήσαμε ε, να περιγράψουμε όσο γίνεται καλύτερα το εργαλείο αυτό ε, με, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εν συντομία δηλαδή προσπαθήσαμε το εργαλείο αυτό να ε, αντικατοπτρίζει τις βασικές αρχές ε, αλλά και τις ε, προοπτικές επί των οποίων συμφωνήσαμε και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη και στα πλαίσια του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και, που, και σαν κράτη-μέλη και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προσυπογράψει ως στόχους που αξίζει να προασπίσει κανείς. Επίσης, τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης απόφασης είναι σημαντικά. Τροποποίησαμε το κείμενο της Κομισιόν, έτσι ώστε η διαφάνεια να είναι μεγαλύτερη. Ο, να υπάρχει μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ε, πάντα προσπαθώντας να γίνει σεβαστή η αρχή της συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών θα βρείτε στις ε, πολλές τροπολογίες μας, ε, αυτές που υποβάλαμε για το κείμενο αυτό, κυρίως ε, για το άρθρο 34β, τροπολογία 238, που αποσκοπεί σε μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου μέσα από ενισχυμένο διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο αφενός, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν Αφετέρου. Αυτό είναι ένα μέρος της προσπάθειας βελτίωσης. Το άλλο αφορά τη βελτίωση της θέσης μας όσον αφορά την ε, συναπόφαση σε θέματα εμπλοκής ε, στο σύστημα. Και εδώ οδηγηθήκαμε από, την, ε, από το εξής ερώτημα. Τι είναι καλό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όμως δεν θα ενοχλεί και παρεμποδίζει την υλοποίηση αυτών των εργαλείων. Τα καταφέραμε νομίζω προσπαθώντας να, συζητήσουμε, να συζητούμε ταυτόχρονα και παράλληλα και με την ε, Κομισιόν έτσι ώστε πραγματικά να βρούμε τρόπο για βελτίωση ουσιαστική της θέσης του Κοινοβουλίου. Οφείλω να ομολογήσω ότι η Κομισιόν, την οποία ευχαριστώ για την ε, μεγάλη διαθεσιμότητα, ε, δεν μας ε, ενθάρρυνε προς την κατεύθυνση των κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, νομίζω ότι η αντίδραση του Φέλιξ ε, δείχνει ότι καθόλου δεν απομακρύνθηκα από την ε, πραγματικότητα και την αλήθεια, αλλά αυτή είναι και η όρη του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε, δεν ξέρω αν το καταφέραμε πλήρως, άρα προσπαθήσαμε στα πλαίσια ενός επικοδομητικού διαλόγου να δώσουμε στην Κομισιόν να καταλάβει, και νομίζω ότι το κατάλαβε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί πλέον να αρκείται στο status quo Λίγες είναι οι προτάσει βελτίωση, βελτίωσης, αλλά είναι ουσιαστικέ. Έχουμε εισαγάγει 8 κατεξουσιοδότηση πράξης, γιατί θα πρέπει να έχει λόγο και το Κοινοβούλιο στις διαδικασίες αυτές. Για μία ακόμα φορά δεν προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε την Κομισιόν ή την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις, ε, ε, στην εργασία τους. Αντιθέτως, θέλουμε να μπορούμε να έχουμε λόγο όσον αφορά ε, μεγάλες στρατηγικές οι οποίες απαιτούν και μεγάλη υψηλή χρηματοδότηση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ούτως ή άλλως πρέπει να εξηγηθούν τα πράγματα στους ε, βουλευτές ξανά και ξανά ε, γιατί είναι λίγοι οι παρόντες και επομένως στις ερχόμενες εβδομάδες θα πρέπει πολλούς να ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πρέντα, εκ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα πω δύο λόγια για την εργασία που κάναμε για τις διάφορες πολιτικές. Θα ξεκινήσω με τη γειτονία. Και θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι εκφράσαμε μια θέση στο Κοινοβούλιο για ανάγκη χωριστού εργαλείου και λυπούμε που η Κομισιόν δεν ενστερνίστηκε αυτήν την ε, βούληση για ξεχωριστό εργαλείο. Επίσης, στην ετολογική σκέψη ανέφερα ε, ότι είμαστε ανοιχτοί για περαιτέρω ε, διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για το ενδεχόμενο αυτού του ξεχωρίσματος λοιπόν ε, του εργαλείου ε, και του μηχανισμού για την ε, γειτονία, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις χώρες γειτονίας Ανατολής, Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης. Εγώ είπα επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να βάζουμε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο τη Γεωργία με τη Βολιβία, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη διάρθρωση αυτού του ε, εργαλείου. Προς ώρας πάντως θεωρώ ότι έχουμε δουλέψει με αποτελεσματικότητα και με αίσθημα ευθύνης έτσι ώστε να βελτιώσουμε πραγματικά την κατάσταση. Πρέπει να ληφθούν ε, ιδιαίτερα υπόψη ε, οι χώρες της γειτονίας. Προτείνω να ενισχυθούν οι πολιτικές, να υπάρχει στοχευμένη modular προσέγγιση στην πολιτική γειτονία. Όσον αφορά τη σταθερότητα και την ειρήνη, συμφωνούμε να εντάξουμε διατάξεις σε όλους τους πυλώνες, κυρίως πρόληψη των ε, ε, συγκρούσεων ε, και επίσης να αναφερθούμε σε πολιτικές οι οποίες οδηγούν στη σταθερότητα και την ειρήνη. Δύο δις ευρώ για τη σταθεροποίηση στον πυλώνα της άμεσης αντίδρασης. Επίσης βοήθεια για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στις χώρες μέσω χρηματοδότησης του εργαλείου για την ειρήνη. Επίσης, βιώσιμη ανάπτυξη οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν εμείς να ε, χρηματοδοτήσουμε την αγορά ας πούμε εξοπλισμών ή ε, ε, και πυρομαχικών, ε, αντιθέτω, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι χρηματοδοτούμε. Όσον αφορά ε, τι ε, χώρε ενδιάμεσου εισοδήματο και τι βιομηχανοποιημένε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει καλή συνεργασία με τι χώρε ε, ενδιάμεσου επίπεδου, έτσι ώστε να υπάρχει δι, ε, ε, αμφίδρομη σχέση. Επίση, προτείνουμε το πρόγραμμα για την εξωτερική πολιτική να, γίνει θεματικό πρόγραμμα. Αυτά με δύο λόγια αλλά θα ήθελα στο τέλος της παρέμβασής μου να ευχαριστήσω την Γραμματεία και των δύο κοινοβουλευτικών μας επιτροπών, διότι δούλεψαν με εξαιρετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματι το προσωπικό μας δήλωψε σκληρά. Είναι πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις συνεισηγητές από δύο επιτροπές και μάλιστα όλα αυτά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ο Φρανκ Έγγελ από το ΕΛΚ της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Θα αρχίσω ακριβώς εκεί που σταμάτησε ο Κριστιαν. Δηλαδή και εγώ ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και από το προσωπικό και από την ομάδα και από τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές που επιτέλεσαν ένα πάρα πολύ αξιόλογο έργο για να καταλήξουμε σε αυτές τις 200 περίπου σελίδες και 400 περίπου τροπολογίες. Γιγάντιο έργο. Τα εξής θέλω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας. Θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε ότι δεν έχουμε έναν ενίο μηχανισμό, ούτε δύο, ούτε ένα μηχανισμό για την ανάπτυξη, αν δεν καταφέρουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης να αποτελεί μέρος του προπολογισμού, κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι κεκτημένο στο Συμβούλιο. Και φαίνεται ότι όλο και κάποια χώρα μέλος, και μάλιστα μεγάλη κάποια, δεν φαίνεται να συμφωνεί. Οπότε όλα αυτά που κάνουμε και όλα αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαρτηθούν από αυτό, από το να μπει στο προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Τώρα, τι κάναμε εμείς ως συνεισηγητές για την ε, υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα. Προβλέψαμε κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για κάποια πράγματα που θέλουμε να ελοπιθούν. Η μεγάλη στρατηγική για την Αφρική πρώτα απ' όλα, η εταιρική σχέση Ευρώπης-Αφρικής, που σήμερα έτσι όπως γεωγραφικά κατανέμεται η εξωτερική βοήθεια δεν είναι σαφές, ενώ η Αφρική σήμερα ακόμα είναι σαφές ότι αποτελείται από μια περιοχή που θεωρείται γειτονίας γιατί βρίσκεται κοντά σε εμά και από μια άλλη που είναι η ποσαχάρια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να βρούμε σημεία σύνδεσης και με συγκεκριμένη χρηματοδότηση μιας πολιτικής που να απευθύνεται στο σύνολο της Αφρικανικής Υπήρου και έτσι να έχουμε μια πραγματικά εταιρική σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο. Το ίδιο ισχύει και για μια άλλη γεωγραφική περιοχή ε, στις χώρες ΣΑΚΕ. Τώρα έχουμε μια γεωγραφική κατανομή της εξωτερικής δράσης που χωρίζει την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Αν λοιπόν διατηρήσουμε την εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ, δεν είναι μια ιδανική κατάσταση αυτή θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη πραγματικότητα για τη χρηματοδότηση των χωρών και στο μέλλον. Ο Σάρλ αναφέρθηκε στη διακυβέρνηση και τον προγραμματισμό που θα είναι πιο θετικό. Αυτό έχει να κάνει και με τι αναπτυσσόμενες χώρε Και χαίρομαι γι' αυτό. Αν κάναμε αυτό που προτείνει ο εισηγητής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βαρύνει περισσότερο στους συγκεκριμένους προσανατολισμούς αναχώρα ή και αναπεριφέρεια στην πολιτική μας συνεργασία με την Αφρική. Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποτελούσε ένα πραγματικό εταίρο για την πολιτική που θα εφαρμόζεται. Η κατάσταση βέβαια δεν είναι ίδια στην κεντρική ε, Αφρική ή τη Μαυριτανία ή την Τανζανία. Και θα ολοκληρώσω με ένα προβληματισμό ο οποίος δεν έχει λυθεί ακόμα και είναι και δύσκολο να λυθεί ποιος είναι ο ρόλος των εταίρων και κυρίως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην υλοποίηση της πολιτικής χρηματοδότησης. Κάποιοι κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θέλει να γίνει τράπεζα η ίδια και ότι θέλησε να απομακρύνει την ΕΤΕΠ από τον ρόλο της που είναι ο πρώτος εταίρος για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης. Ενώ η ΕΤΕΠ σήμερα ένα πολύ περιορισμένο ποσοστό του συνολικού ποσού που απευθύνεται στην αναπτυξιακή βοήθεια πηγαίνει στην Αφρική. Ενώ η Επιτροπή, απ' την άλλη, δεν σκοπεύει να γίνει τράπεζα. Ίσως όμως ήρθε η ώρα να καθίσουμε να σκεφτούμε και με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με την ΕΤΕΠ μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, Ανάπτυξης, Αναπτυξιακή Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η ΕΤΕΠ, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε ίσως να αποκτήσει στο μέλλον ένα σκέλος που να ασχολείται με την ανάπτυξη ή να έχουμε μια καθαρά Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εκτός ΕΤΕΠ. Θα έπρεπε να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να έχουν όλοι οι ευρωπαϊκέ Αναπτυξιακές τράπεζε ή Αναπτυξιακές τράπεζε, τέλο πάντων υπάρχουν σε όλες τις χώρες ε, στην Αφρική υπάρχει, στην Ασία υπάρχει, στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τέτοια. Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό μακροπρόθεσμα. Αυτό θα πρέπει να το λύσουμε. Μπορούμε λοιπόν να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε Φρανκ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Παντσέρη από την Υποτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, ε, ε, γιατί πραγματικά η συνεργασία ήταν καλύτερα. Εγώ είχα το καλύτερο κομμάτι της ε, έκθεσης. Χαίρομαι γι' αυτό. Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες έχουμε ε, εισάγει κάποιες νέες ε, διατάξεις οι οποίες δίνουν την δυνατότητα ε, να ανακληθεί η υποστήριξη προς μια χώρα σε περίπτωση διαρκούς και επίμονης έλλειψης συμμόρφωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 500 εκατομμύρια ευρώ έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση ε, της κοινωνίας των πολιτών για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, ε, έχουμε 700.000 700.000 ε, ευρώ ε, καθώς επίσης και για μη κυβερνητικές οργανώσεις 0,5. Όσον αφορά το FSD+, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο ε, και ότι θα πρέπει να δοθούν 60 δισευρώ για τις επιχειρήσεις όσον αφορά ε, τις ε, επενδύσεις οι οποίες αφορούν ε, την συμμόρφωση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, της, το περιβάλλον κλπ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται. Επίσης στο βασικό άρθρο και όχι στο κύριο σώμα δηλαδή και όχι στα παραρτήματα έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία αυτά. Επίσης οι ιδέες των συνεισηγητών ε, είναι και οι απόψει του είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν οι αρχέ έτσι ώστε να υπάρξει δημοκρατικό έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα να αφήνεται και χώρο για ευελιξία και, διακριτική ε, δυνατότητα ε, των χωρών να κινηθούν με τις δικές τους ε, δυνάμεις. Θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να υπάρξουν και τροπολογίες ε, οι οποίες καλύτερα να αναφέρονται εις, ε, την, στις θεματικές και γεωγραφικές ισορροπίες και τέλος μέσω της εκθέσεως επαναλαμβάνουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να δοθούν 3,5 δις στην Αφρική 2,4 στην υποσαχάρια και 1,1 ε, ε, στο εργαλείο για την Αφρική. Αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις συνεισηγητές με τους οποίους ε, συνεργαστήκαμε σωστά νομίζω και καλά τους τελευταίους τρεις μήνες έτσι ώστε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα καλό συνολικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έπρεπε να πω ότι ο κύριος Παντζέρη, εκτός από πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι και ο τέταρτος συνεισηγητής ε, εκ μέρους των σοσιαλιστών. Λοιπόν, να δούμε τους σκιώδεις. Ε, θα σας πω τα ονόματα που έχω, ε, τα ονόματα αγορατών, αγορητών. I've got Sabine Michael and Edward Does anybody else... Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο για να του δώσουμε τον αντίστοιχο χρόνο αγόρευσης. Όχι. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτούς τους τέσσερις ομιλητές και την Κομισιόν αμέσως μετά. Κύριος Αστροβίσιος. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την κυρία Μαρσεσάκια η οποία συγχαίρει τους συνσηγητές για το σκληρό έργο τους που επιτέλεσαν τις τελευταίες ε, εβδομάδες. Το γεγονός ότι οι ίδιοι συνεισηγητές έχουν ε, καταθέσει πάνω από 300 τροπολογίες ε, καταδεικνύει και την πυροπλοκότητα του θέματος. Ελπίζει ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο πριν την εκνοή της θητείας. Σημαντικό όμως είναι ε, αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε στην, ε, σε μια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα τη χάνει τη υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Θα υποβάλει συγκεκριμένε τροπολογίε που θα επικεντρώνονται στα εξή. Πρώτον, στο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει σαφή οριζόντια δομή διακυβέρνηση ε, και που θα καλύπτει την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η οποία θα λογοδοτεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, πρέπει να τεθούν τα ανθρωπίνα δικαιώματα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξωτερικών σχέσεων. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει σαφές πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο υπό το οποίο μπορούν να αναπτύσσονται προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης. Και τέταρτον, να υπάρχουν σαφείς δείκτες για κάθε δράση καθώς και αξιολόγηση σε τακτική βάση. Εκ μέρου της Μαρίσια Σάκε θέλω να ευχηθώ ε, κάθε επιτυχία στους συνεισηγητές. Θα παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά, ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό και ισχυρό κείμενο στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λόζινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά θέλω να τονίσω ότι η ομάδα μου και εγώ ανησυχούμε πολύ για το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κονδύλια τα οποία κατευθύνονται ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια υπό το άρθρο 287 της συνθήκης που ορίζει ότι στόχος είναι η καταπολέμηση του αποκλεισμού και της, ευτι... και της φτώχειας πλέον ε, αξιοποιούνται για την μετανάστευση ή ακόμη και για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό ε, συνέβη και στο μηχανισμό για τη σταθερότητα και την ειρήνη αλλά και στα Trust Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική και αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με την συγχώνευση του, των ταμείων του NDICI. Γι' αυτό χαιρετίζω το γεγονός ότι οι συνεισηγητές έχουν υποβάλει τροπολογίες για την ενίσχυση ε, του άρθρου 287 ε, και για το, ότι, ότι έχουν επιλέξει μια άλλη διατύπωση για τη μετανάστευση, όπου μιλούν πλέον για αναγκαστική μετανάστευση. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι η συγχώνευση αυτών των ταμείων και των χρηματοδοτικών μέσων δεν θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά σε μεγαλύτερη αδιαφάνεια. Κατά τη γνώμη μας, η συγχώνευση όλων αυτών των τομέων πολιτικής στο νέο NDICI συμπεριλαμβανομένη τη αναπτυξιακή βοήθεια, τελικά θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των ε, διαφόρων τομέων πολιτική και την υπαγωγή τους στα καθαρά γεωπολιτικά οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι ε, ουσιώδη συνεισφορά στη σταθερότητα και την ειρήνη. Έχω να απευθύνω και ένα ερώτημα ιδίως στον κύριο Πρέντα ως ε, υπευθύνου για το θέμα αυτό από πλευράς ΑΦΕΤ. Είπατε στην τελευταία ε, συνάντηση των σκιωδών ότι σε κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις που είχατε με την Κομισιόν προσπαθήσατε σύμφωνα με την απόφαση ε, της ε, ΑΦΕΤ ότι το, ο μηχανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έχει αυτόνομο, ανεξάρτητο χαρακτήρα. Βεβαίως δεν ήταν ευήκοα τα ότα που άκουσαν αυτήν την, την πρότασή σας τι σας έκανε να αλλάξετε γνώμη. Διότι βλέπω ότι πλέον τα δύο αυτά εργαλεία ε, βρίσκονται εντός του NCICI. Εγώ επαναλαμβάνω εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας ότι θεωρούμε ότι είναι λάθος η συγχώνευση όλων αυτών των μηχανισμών και των εργαλείων γιατί θα οδηγήσει και μεταξύ άλλων σε ε, ε πιο δύσκολο, θα καταστήσει πιο δύσκολο το έργο ε, ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη οι κατεξοδότηση πράξεις που διέπουν τα ξεχωριστά εργαλεία έχουμε δει ότι οδήγησαν σε μικρότερη λογοδοσία ε, απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αυτό θα αλλάξει τώρα που θα συγχωνευτούν μάλιστα τα εργαλεία. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει στο, ελάχιστο, στο μέτρο του ελάχιστου δυνατού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατεξοδότηση ε, πράξεις. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον ενισχυμένο διάλογο και τον στρατηγικό διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ερωτήσεις για τους συνεισηγητές μας και να δώσουμε το λόγο στους άλλους ομιλητές που δεν είναι σκιώδεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Μιχαήλ Γκάλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές και να τους διαβεβαιώσω ότι η κριτική που θα ασκήσω δεν απευθύνεται στους ίδιους προσωπικά, αλλά στη διαδικασία που επελέγει. Διότι ε, πραγματικά έχω σοβαρές επιφυλάξεις ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί, θεωρώ ότι δεν επαρκεί για αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο έργο που έχουμε μπροστά μας. Δεν ε, συμβάλλουμε στο να γίνει ουσιαστική δουλειά στις επιτροπές μας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε από ανταλλαγή απόψεων ε, και εξέταση των θεμάτων αυτών, ούτε μας, ε, ούτε μας αρκεί ο χρόνος για να δούμε διάφορες διαστάσεις και αποχρώσεις των, του θέματος αυτού. Είπαν, είπα και ο κύριος ε, Γκέρν σήμερα ότι έχουμε περισσότερους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων σήμερα εδώ στην αίθουσα παρά ευρωβουλευτές. είναι χαρακτηριστικό. Εγώ θα ήθελα να είχαμε ακολουθήσει τη διαδικασία που είχαμε ακολουθήσει το 2006, η οποία ήταν πολύ πιο αποτελεσματική. Εγώ είμαι από τους λίγους που έχει, έχουν εργαστεί ε, στους ε, αρμόδιους ε, φορείς, στις αρμόδιες επιτροπές τα τελευταία 20 χρόνια, στις ΕΝΤΕ, στην ΤΕΒΕ, στην ΑΦΕΤ, σε διάφορες αντιπροσωπείες για εταιρικές σχέσεις με χώρες του Νότου, του Βορρά. Σήμερα μάλιστα ήρθα και από την Τουρκία. Για μένα σημαντικό είναι ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός και εφαρμόσιμος. Γι' αυτό και θέλω να αναφερθώ σε τρία ουσιώδη θέματα που με απασχολούν. Έχω πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά συγκεκριμένε ε, δεσμεύσει κονδυλίων. Σωστά διάβασα, το 95% των δαπανών θα κατευθύνονται σε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ποια μέτρα εξωτερικής πολιτικής λοιπόν θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από αυτό το μηχανισμό και ενώ ολόκληρο το εύρος της εξωτερικής συνδρομής βοήθειας και της εξωτερικής συνεργασίας. Θέλω με όλα τα πιθανά μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατανομή των μέτρων αυτών, πώς ακριβώς τελικά αυτά θα, θα πέφτουν στο κάθε μηχανισμό. Δεύτερον, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και με περιφέρειες τρίτων χωρών, θα πρέπει αυτά τα μέτρα να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται και στην πράξη, στην εφαρμογή της, πολιτικής, ε, ε, της εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να οδηγήσουν και σε αλλαγή των, κειμένων, των μας. Δεν θα πρέπει οι νομικές πράξεις που εγκρίνουμε να δίνουν τη δυνατότητα και στους ευρωβουλευτές να ε, υπηρετούν αυτούς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα. Ποιο είναι το όφελος από τη συγχώνευση αυτών των 7 αυτόνομων εργαλείων σε ένα και ποια είναι τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή την απόφαση. Και τέλος, ε, για τον, ένα αυτόνομο εργαλείο θα μπορούσε να, να χρηματοδοτηθεί και να δημιουργηθεί για τον τομέα της δημοκρατίας και των εκλογών. Εδώ έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή είναι μια διαδικασία εξαιρετικά ε, δύσκολη και επίπονη σε χώρες μετάβασης, σε χώρες αναπτυσσόμενες. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι θα πρέπει στο μέλλον να προσφέρει θεσμικά και χρηματοδοτικά μέσα στήριξης και βοήθειας σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και να προβλέπονται και στη δική μας εργαλειοθήκη. <coughs> Πρόεδρος. 92% είναι το ODA για τις λιγότερο αναπτυγμένες και την αναπτυξιακή βοήθεια. Και ο συγητής λέει να είναι 95%. Μπορεί να το εξηγήσει όμως. Edward Κούκαν είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τους συγητές, συνεισηγητές και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κειμένου αυτού. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Είδα την πρώτη πρόταση της Επιτροπής. Εγώ ήμουνα εισηγητής νωρίτερα και είδα ότι είναι ενδιαφέρον να βάλουμε κάτω από μέσα σε ένα πλαίσιο μάλλον όλη την εξωτερική βοήθεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον, τη βασική φιλοσοφία του Μηχανισμού Γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές σχέσεις στη γειτονία μας, αλλά καλό είναι να υπογραμμίσουμε τη συνεργασία μας και να ακολουθούμε λύσεις καλά προσαρμοσμένες στην κάθε περίπτωση για τις γείτονες χώρες. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης περισσότερη προβολή για την ευρωπαϊκή βοήθεια και σύγκληση των ευρωπαϊκών μας στόχων στην περιοχή. Θα ήθελα να δω επίσης την εγγύηση. Ο προϋπολογισμός στο μηχανισμό αυτό να προσανατολίζεται στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στόχους των χωρών αυτών και όχι τόσο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, συμφωνώ με την αρχή περισσότερα για περισσότερα. Και αυτό πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα στους γειτονές μας. Να ανταμείβουμε αυτούς οι οποίοι στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικονομικής ε, διακυβέρνησης μέσω μεταρρυθμίσεων. Συγχρόνως, οι χώρες στη γειτονία μας πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις σχέσεις που έχουμε με την κάθε χώρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τις χώρες που έχουν συμφωνία σύνδεσης μαζί μας. Πρέπει να βρούμε και το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητήσουμε τις επιδόσεις στα πλαίσια του περισσότερα για περισσότερα. Ο στρατηγικός διάλογος δεν έχει ικανοποιήσει τους στόχους μας. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερο διαρθρωμένο πλαίσιο για διάλογο. Τέλος, όσον αφορά το EFS-SYN, πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι περιλαμβάνει ο μηχανισμός αυτός. Και να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα πρέπει να τονίζει τους στόχους μας και τις αρχές μας στην εκάστοτε περιοχή. Και το EFSD και το ECI ε, θα πρέπει να κάνουν την πολιτική μας να διέπεται από περισσότερη συνοχή. Μιλάμε για οικονομικούς μηχανισμούς. Πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το ρόλο των ε, ε, οικονομικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνει ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα σχεδιάζεται η οικονομική μας αρρωγή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε στον Πενάν συνάντηση και πολλοί συνάδελφοι είναι εκεί και γι' αυτό δεν είναι εδώ. Γι' αυτό είμαστε λίγοι. Ο κύριος Αστροβίτσιος είναι επόμενος. Μιλάει εκ μέρους του αυτού του αυτή τη φορά. Έχω εντολή, έχω φωνή, οπότε μπορώ να μιλήσω, λέει ο κύριος Αστροβίτσιος. Μιλάμε για τη συγχώνευση ε, διάφορων μηχανισμών σε κάτι νέο. Αυτό το νέο λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό και πλήρες. Κατά τη γνώμη μου όμως, όταν κοιτάω την τροποποιητική διαδικασία, λέω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προηγούμενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχήν. Να μην υπάρχει άρση της βοήθειας άπαξ και τα κονδύλια διοχετεύονται ως πράξη φιλίας χωρίς να ζητάμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η οικονομική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διοχετεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη προβολή της αρρωγής μας στις ε, διαφερόμενες χώρες, το παν αυτό. Δεύτερον, να υπάρχει μια ρήτρα ασφαλείας για να μην καταλήγουμε να πετάμε τα χρήματά μας σε δικτατορίες και αυταρχικά καθεστώτα. Και έχουμε αρκετά στον κόσμο τέτοια. Και τρίτον, να αποτελούν στοιχείο πίεσης απέναντι σε τρίτες χώρες για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας υπέρ της ε, δικιάς μας ασφάλειας. Είμαι υπέρ επίσης της παύσης ε, αρρωγής, της αιρεσιμότητας που θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως όρος στο μηχανισμό αυτόν. Χαίρομαι για το άρθρο 15α λοιπόν που μιλάει για την παύση αρρωγής. Εφόσον δεν τηρούνται οι αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, τότε θα έπρεπε να προχωρούμε σε πάυση της αρρωγής. Ε, κάτι που ψηφίσαμε στη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ ήταν ε, το κείμενο για την πυρηνική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το μηχανισμό αυτόν ε, στηρίζει ότι η βοήθειά μας θα εξαρτάται από την πρόσφατη συνεργασία μας και το άνοιγμα στα πυρηνικά, κυρίως όταν υπάρχουν υπόνοιες στην ε, γειτονία μας. Όταν δηλαδή έχουμε αμφιβολίες για την ασφάλεια των πυρηνικών σε κάποιες ε, χώρες στη γειτονιά μας. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να συμπληρωθεί στην αιρεσιμότητα που αναφέραμε πριν. Όταν υπάρχει κάποια παραβίαση στις δημοκρατικές αρχές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έτσι ολοκληρώνω το κατάλογο των Ευρωβουλευτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει τον λόγο τώρα. Γενικός Γραμματέας τη ΤΕΦΚΟ και Γειτονίας, Στεφάνο Μοντσοβίση, ΤΕΦΚΟ. Δύο λεπτά θα έχετε ο καθένας, να ξέρετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και κυρίως βεβαίως τους εισηγητές για την κοινή προσπάθεια που κατέβαλαν ε, για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Προτείνουν ε, κάποιες ε, τροποποιήσεις και η διαδικασία είναι αργή. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το DCI ε, ε, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δοθεί του Κοινοβουλίου, να ενταθεί ο λόγος του Κοινοβουλίου στα πλαίσια ε, της παρουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Πρέπει να δούμε λίγο βέβαια τα γενικά στοιχεία της διάρθρωσης, γιατί θα έχουμε και άλλες φορές την ευκαιρία και την δυνατότητα να μιλήσουμε εν λεπτομερία. Τα γενικότερα η ενότητα του εργαλείου ε, είναι ε, ακριβώς το στοιχείο το οποίο ε, είναι πολύ θετικό. Να μην λησμονούμε όμως ότι το εργαλείο δεν είναι η πολιτική. Μέσω των εργαλείων γίνεται η πολιτική. Επίσης, στενή συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, ε, ε, αμέσως μετά έρχεται η διακυβέρνηση. Αυτό το κατανοούμε απολύτω και βεβαίω θέλουμε να το προσυπογράψουμε. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι σύμφωνα και με τις Γενικές Αρχές του Κοινοβουλίου, η κύρια απάντηση από εσά ήταν η κατεξουσιοδότηση πράξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ούτε εγώ, αλλά γενικότερα ως ε, ε, ε, υπηρεσία δεν είμαστε πεπισμένοι ε, για, την, ε, το εργαλείο αυτό. Πρώτον, τίθεται ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας. Ε, δεν συμμορφούνται αυτό με την αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, και δύσκολο να καταλάβουμε, σύμφωνα και με την, τις εξουσιοδότηση πράξης, είναι οι διαφορές μπορούν να προκύψουν. Τέλος, μπορεί ο αντίκτυπος να είναι διαφοροποιημένος στο κοινό πρόγραμμα. Επομένως, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε με τη διακυβέρνηση από ελαφρώς διαφορετική σκοπιά. σκοπιά. Όλοι βεβαίως συμφωνούμε ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο στην ε, διαμόρφωση πολιτικών εξωτερικής δράσης. Αυτό όμως θα πρέπει να ξεχωριστεί από ε, έναν έλεγχο τύπου scrutiny control για τα μικροοικονομικά. Θα πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά έχοντας αδεδομένο ότι η διακυβέρνηση είναι μια μια ισχυρή θέση. Δεύτερον, όσον ε, αφορά ε, ε, την ε, ε, αναπτυξιακή πορεία. Ε, ε χαιρόμαστε. Ας μην λησμονούμε ότι το εργαλείο αυτό αντικαθιστά μια σειρά από άλλα εργαλεία τα οποία δεν είχαν απολύτως τον ίδιο στόχο και ότι εν πάση περιπτώσει έχει ήδη αποδειχθεί η, η πραγματική αξία, προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα θέματα. Το 95% ίσως ε, δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ε, για το χρηματοδοτικό ε, στοιχείο ε, ε, ενδεχομένως ε, διαφορετική ρήτρα κατανομής, κλίδα κατανομής, ίσως δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όντως το κεκτημένο, όπως είπατε και με, μερικοί μεταξύ ημών. Θα πρέπει ίσως λοιπόν να πούμε πώ είναι δυνατόν με μεγαλύτερη διαφάνεια τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το τελευταίο σχεδόν σημείο μου είναι το θέμα των επενδύσεων. Είναι σαφές ότι δεν θέλουμε το εργαλείο αυτό να είναι τράπεζα, Θέλουμε όμως ε, να ε, ταυτιστεί, να ευθυγραμμιστεί μάλλον με, την, ε, με το θεματολόγιο για την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, εδώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει σημαντικό επενδυτικό ρόλο, αλλά έχει και ανοιχτή αρχιτεκτονική, γιατί υπάρχουν πολλές αναπτυξιακές τράπεζες στις χώρες και επομένως εδώ θέλουμε να ενισχυθεί ο κοινός προγραμματισμός ε, πάντως ε, συμφωνούμε με πολλά από τα στοιχεία τα οποία αναφέρετε. Τέλος, ε, το λέω εξ ονόματος όλων, σημαντικότερο, ισχυρότερο ρόλο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Κοιτάξτε, μαζί διαχειριζόμαστε, μαζί δουλεύουμε. Νομίζω ότι ε, ήδη στην απόφαση ε, που θεσπίζει την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, δίνει συγκεκριμένο ρόλο στην υπηρεσία όσον αφορά την ηγεσία από πολιτικής απόψεως. Βεβαίως θέλουμε να δουλέψουμε από κοινού, αλλά στην ουσία εμείς κάνουμε αυτό που έχουμε δεσμευτεί εξ αρχής να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεπεράσατε το χρόνο σας, αλλά ήταν σημαντικό το θέμα. Έχουμε μαζί μας και τον Γενικό Διευθυντή της DGNIR, ο κύριος Ντάνιελσον. Ευχαριστώ που μου υπενθυμίσατε ότι μας πιέζει ο χρόνος, άρα λιγότερος χρόνος για μένα. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεισηγητές, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι ομιλητές, που θεωρούμε ότι τροφοδοτεί τη συζήτησή μας με επικοδομητικό τρόπο για το μηχανισμό γειτονία και το νέο ενιαίο μηχανισμό που θεσπίζεται. Θέλω να τονίσω τη σημασία που αποδίδουμε σε αυτόν τον μηχανισμό από άποψη της πολιτικής γειτονίας και αυτό το λέω διότι ο μηχανισμός αυτός προσφέρει ευελιξία, απλούστευση των κανόνων και μας εξοπλίζει καλύτερα για να εργαστούμε επί όλων αυτών που ανέφερε ο κύριος Κούκαν όσον αφορά τις ε, ιδιαιτερότητες που έχει η συνεργασία μας με τους εταίρους της γειτονίας. Και αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουμε ότι αυτός ο νέος μηχανισμός είναι ε, ο σωστός τρόπος προσέγγισης για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δράση και την ευρωπαϊκή στήριξη ε, για τις διάφορες μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες επιδιώκουμε οι εταίροι μας να υλοποιήσουν. Αυτό είναι το πρώτο μας σχόλιο. Δεύτερον, χαιρετίζουμε ε, θερμά αυτά που αναφέρει η έκθεση σχετικά με την σημασία των επιδόσεων. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο για τις παρεμβάσεις μας στην γειτονία. Νομίζω ότι οι συγητές ορθώς το διατυπώνουν. Ε, το πώς θα βελτιωθεί αυτή η παρέμβασή μας βεβαίως μπορούμε να το συζητήσουμε αλλά να θυμόμαστε πάντοτε ότι δεν θα πρέπει να βρεθούμε σε θέση όπου θα είναι πραγματικά πιο δύσκολο να έχουμε ε, επιρροή όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκουμε να γίνουν στις χώρες που στηρίζουμε. Τέλο, όσον αφορά την προβολή και την ορατότητα, θεωρώ ότι αυτό ο μηχανισμό, ο ενιαίο, θα μα δώσει τη δυνατότητα να προβάλλουμε καλύτερα το έργο μα, γιατί θα είναι πλέον σαφέ στου εταίρου μα πώ εργαζόμαστε και μέσω ποιου μηχανισμού. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να, κατα... να, να εγκριθεί, να θεσπιστεί ένας τέτοιος ενιαίος μηχανισμός, ο οποίος πραγματικά θεωρώ ότι θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προβολή και την ορατότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Κρίστιαν Λέφλερ. Δεν ξέρω πού είναι. Α, σας βλέπω, ναι. Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ναι, κυρία ε, Πρόεδρε, κρυβόμουν λίγο. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και να επαναλάβω και εγώ ε, τις ευχαριστίες των ε, προλαλισσάντων προς τους συνεισηγητές για το εξαιρετικό τους έργο. την ξεκάθαρη παρουσίαση των θέσεών τους και τις συστάσεις στις οποίες έχουν καταλήξει. Θεωρώ ότι η ετοιμότητα που αναδίδεται μέσα από την έκθεση για την ε, συνεργασία, για την ε, προώθηση της ε, εξωτερικής παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα στοιχείο πολύ ενθαρρυντικό για εμάς. Ο κύριος Πρέντα εξέφρασε κάποιες προσωπικές ε, αμφιβολίες όσον αφορά την συγχώνευση όλων των μηχανισμών σε ένα εργαλείο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την ε, Γεωργία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη Βολιβία, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Βολιβία σε σχέση με την Νορβηγία ή τον Καναδά. Το σημαντικό είναι ότι ο μηχανισμός αυτός ο νέος, ο ενιαίο μας δίνει την ευελιξία ώστε σε διαφορετικές, να ακολουθούμε διαφορετικές προσεγγίσεις κατά θεματικό τρόπο ή και κατά γεωγραφική περιοχή στις ε, παρεμβάσεις μας και στη συνεργασία μας. Και αυτό είναι και ο λόγος που ο μηχανισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενσωματώνεται πλέον στον νέο μηχανισμό. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα περιφερειακό ζήτημα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελεί βασικό στοιχείο της εξωτερικής μας παρέμβασης ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφού λοιπόν είναι βασικό συστατικό στοιχείο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις μας, σε όλες τις παραμβάσει μας. Και γι' αυτό το λόγο συγχωνεύουμε και ο μηχανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτόν τον νέο ενιαίο μηχανισμό, ε, λαμβάνοντας πλέον υπόψη αυτήν τη διάσταση στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε όλες τις ε, παρεμβάσεις μας. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε ο, η συγχώνευση αυτή και αυτό ανέφερε και ο Στέφανο σε σχέση με την συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες για, ένα, για την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων για να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργούμε στην ουσία ένα ενιαίο συνεκτικό πλαίσιο μέσω αυτού του μηχανισμού για να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική δυναμική για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Για να το κάνουμε αυτό, για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται ενισχυμένος πολιτικός διάλογος. Και αυτό είναι βασικό στοιχείο για τη διακυβέρνηση του μηχανισμού. Ο κ. Μασκεβίζη ε, ανέφερε ότι αυτός ο διάλογος θα ε, πηγαίνει και από τα κάτω προς τα πάνω και από τα πάνω όμως προς τα κάτω. Όπως ανέφερε και ο κύριος Αστροβίζιος, και αυτό αφορά και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε όλες τις φάσεις. Και πρέπει επίσης να πω ότι θα πρέπει να γίνεται και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων. Όχι μόνο πριν την κατάρτισή τους ή μετά εκ των υστέρων, αλλά θα πρέπει να είναι ένα βασικό διαρκές στοιχείο το οποίο θα μας ε, δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πολιτική καθοδήγηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από, το, από τα κράτη-μέλη για το πώς θα συνεχίσουμε και θα υλοποιούμε αυτή την ε, πολιτική, τα προγράμματά μας. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία που εκφράζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για, την, για τις κατεξιότητες πράξεις. Εγώ ειχαμε μετρήσει 7, ο κύριος Γκιόρεντς με διόρθωσε και μου είπε ότι είναι 8. Θα υπάρχουν λοιπόν εξοδότηση πράξεις, αλλά ε, δεν θεωρούμε ούτε εμείς ότι ε, είναι το καλύτερο εργαλείο για να εξασφαλιστεί μια δυναμική διακυβέρνηση με πραγματική επικέντρωση στους στόχους που έχουμε θέσει για την επόμενη περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ συνεισηγητές. Δυστυχώς ε, μας τελειώνει ο χρόνος και έχουμε, η ΑΦΕΤ μάλλον διοργανώνει και σημαντική ακρόαση για τη σχέση με, τις ε, με την Ιαπωνία. Θέλω, θέλετε να σας δώσω το, το λόγο. Εντάξει, Σαρ πρώτος, αλλά πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω στις παρατηρήσεις μου τις ευχαριστίες στις ομάδες που μας στήριξαν, είτε πρόκειται για μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, είτε της Επιτροπής Ανάπτυξης. Και θέλω να προσθέσω και κάτι για μια παρεξήγηση που υπάρχει ανάμεσα στις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Εμείς δεν είμαστε φετιχιστές με τις πράξεις. Ξέρω ότι πολλοί υποβάλλουν τέτοιε. Και ο τέο επίτροπο, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου που γνωρίζει πολύ καλά και εκείνο υπέβαλε τροπολογίε. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε τόσο μακριά όσο ο πρόεδρος μας. Είπαμε ότι είμαστε ένα κοινοβουλευτικό σώμα με τα προνομιά του. Στην αρχή είμαστε περισσότερο ένας ακαδημαϊκός χώρος για αυτούς που γνώρισαν το 1979 1984 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρουν ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα στα περίπρεο υπολογισμού και αγωνιστήκαμε. Και κάθε φορά είχαμε την ίδια αντίδραση. από τη μια αυτή που λέγανε προσοχή, γιατί αν δώσετε δικαιώματα στους ευρωβουλευτές ε, τότε θα χάσετε την ευθύνη. Το αντίθετο έγινε όμως κάθε φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες και τις αναλαμβάνει τις ευθύνες του, δεν τις αποποιείται. Και καταλαβαίνω αυτούς από την Κομισιόν που λένε ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται με τα πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, γνωρίζουμε το ρόλο μας. Αλλά για τις μεγάλες σημαντικές επιλογές δεν μπορεί εμεί να μένουμε στο περιθώριο. Υπάρχει προσφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό, στα πλαίσια ενό ενισχυμένου διαλόγου το λαμβάνουμε υπόψη μας. Αλλά και πάλι είμαστε κάτι παραπάνω από απλούς ακροατές. Ε, δεν δικαιούμαστε απλώς και μόνο ένα briefing. Είμαστε αυτοί που συναποφασίζουν. Και βέβαια και οι χώρες μέλη θέλουν να ακουστεί η δικιά τους φωνή. Και αυτό θα είναι το σημαντικό στις συζητήσεις που θα γίνουν στον τριμερή διάλογο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε επίση είναι να ανταποκριθούμε σε αυτά που ζητάει κοινή γνώμη, η οποία αναρωτιέται τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε χρέος λοιπόν και οφείλουμε να καθησυχάσουμε τους πολίτες για να ξέρει ότι οι άνθρωποι που εξέλεξαν κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους. Όχι για να διαχειριστούν τις δουλειές άλλου, με κάθε σεβασμό το λέω αυτό και προς τον κύριο Λεκλέρ, έχει αλλεργία στον όρο κάτι εξουσιοδότηση πράξης. Μόλις ξεκινάει κανείς ε, με την πρώτη συλλαβή, αμέσως βλέπει την αντίδραση. Μα εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε κάπως τις απόψεις μας. Και πάλι να ξέρετε ότι και οι τέσσερις συνεισηγητές καθίσαμε και συζητήσαμε πολύ σοβαρά για το ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και πιστεύουμε ότι η μέση οδός που επιλέξαμε είναι απόλυτα εφικτή και αποδεκτή θα μπορούσε να είναι και από τα τρία θεσμικά όργανα. Ε, να προσθέσετε κάτι κύριε Πρέντα πολύ σύντομα. Ναι, για να είμαι ευγενή και προ του ε, Ιάπωνε φίλου, οι οποίοι περιμένουν να αρχίσει η ακρόαση που έχουμε προβλέψει για τι σχέσει μα με την Ιαπωνία. Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει ήδη εδώ και 20 λεπτά. Ο κύριος Παντζέρη, έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, εντάξει. Ωραία, οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ τους συνεισηγητές και για την κατεξισοδότηση πράξης. Θέλω να θυμίσω στην Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολλές νομοθετικές προσπάθειες. Ε, πολλές από τις νομοθετικές ε, πράξεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχαν ε, περάσει αν δεν είχατε σύμμαχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Φρόντ για να κλείσει την συνάντηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ όλους τους παρόντες. Οι προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, να ξέρετε. Και στο πνεύμα της κοινή αυτής συνάντησης ε, ζητώ όλες οι ομάδες να φροντίσουν για το συντονισμό των τροπολογιών τους και να φροντίσουν να είναι συνυπογραμμένες από μέλη και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε τις τροπολογίες θα είναι τον Ιανουάριο, 22 Ιανουαρίου. Λίγει λοιπόν αυτό το τμήμα της συνεδρίασης και ο κύριος ε, Φαμπρέντα θα αναλάβει τώρα την Προεδρία για τη συνέχεια.